Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουν έρθει όλοι, όμως ε, θεωρώ πως πρέπει να αρχίσουμε. Διότι έχουμε αρκετά μεγάλες ε, ψηφοφορίες, γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη, με το σημείο 1, την έγκριση δηλαδή της ημερήσιας διάταξης. Εάν συμφωνείτε με το σχέδιο ημερησία διάταξης ή αν υπάρχουν επιθυμίες για να αλλάξει κάτι, να τοποποιηθεί, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε θεωρώ πως εγκρίνεται το σχέδιο ημερησία διάταξης. Δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών από την 21η και 22η Φεβρουαρίου θα βρείτε τα πρακτικά στα έγγραφα που έχετε λάβει. έν υπάρχουν σχόλια, παρατηρήσεις, όχι, δεν υπάρχουν. Τότε λοιπόν προτείνω ως συνήθως να θεωρήσουμε πως τα πρακτικά έχουν εγκριθεί σε ε, αν δεν ε, υπάρχει κάποια αντίρρηση στη διάρκεια της συνεδρίασης. Μετά περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσεις της Προέδρου. Πρώτον, να πω ότι σήμερα υπάρχει διερμηνία στις ακόλουθες γλώσσες γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εσθονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά και ρουμάνικα. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών από τις 19 Μαρτίου 2018, να σας ενημερώσω ότι στις 20 Μαρτίου ε, εστάλησαν με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και δεν υπήρχαν κάποιες ε, ενστάσεις μέχρι τις 22 Μαρτίου, την προθεσμία δηλαδή, επομένως περνάμε στις, στην ενημέρωση για τις ψηφοφορίες. Σήμερα θα ψηφίσουμε δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας, μία νομοθετική γνωμοδότηση και μία έκθεση πρωτοβουλίας. Περνάμε στην έκθεση πρωτοβουλίας εξυγχρονισμός της ε, εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κριστίνα Λουπάτσκα ήταν η συγγήτρια. 485 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό θα έλεγα θέμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω την ε, Κριστίνα εάν ε, θα ήθελε να προσθέσει κάτι, να σχολιάσει κάτι για την έκθεσή της. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πολύ οικοδομητική δουλειά που έχει γίνει για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να, να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές επίσης για την εξαιρετική συνεργασία, καθώς και τους ε, βοηθούς και τη γραμματεία. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τους ε, δικούς μου βοηθούς. Ελπίζω ο τομέας της παιδείας να συνεχίσει να είναι αυτό που μας ενώνει εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα δυνατό μήνυμα που στέλνουμε τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στα κράτη-μέλη με την ε, έκθεση αυτή και θα αρχίσουμε αμέσως. Έχουν αποσυρθεί τροπολογίες 68 και 69, γι' αυτό λοιπόν περνάμε στην συμβαστική τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 96 έχει αποσυρθεί. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται όμως ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 99. Geschlossen. Beides. 13 ψήφοι κατά, 11 υπέρ απορρίπτεται. Λοιπόν, περνάμε στην τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην ΦΕΜ 6, όχι, κατά πίπτη. Η συμβαστική 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 132. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 148. Πέρας. Εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Συμβιβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 και 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 199 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 14 ψήφοι υπέρ 12 κατά εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 224. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 225. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 236. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 246 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 54 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμφιβαστική 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 54 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 296. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 297. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τη 297. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 299. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 300. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 301. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 303. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 304. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 305. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 306. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 307. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 308 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 308 άρχεται η ψηφορία πέρας απορρίπτεται Συμβαστική 58 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φέμ 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 328 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 332 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 64 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Φεμ 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 339 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 343 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 345 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 347 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 357 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 358. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 361. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 362. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 367 έχει αποσυρθεί. 368. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 368. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αποσύρεται και 370, συμβαστική 68, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 374, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 375, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 69, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 380 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ας το ελέγξουμε, αλλά νομίζω πως έχουμε την ίδια πλειοψηφία. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία για την 380. Πέρας. Εγκρίνεται. 13 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. 381 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 70 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 71 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 385 υπέρ, κατά. Αποχές Νομίζω πως εγκρίνεται, ας το ελέγξουμε καλύτερα. 385, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 72, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη 27, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 395 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 398 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 400 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 411. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται. Θα το ελέγξουμε όμως. Δεν σηκώσατε όλοι το χέρι. 411. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 412. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω πως εγκρίνεται. Θα το ελέγξουμε και αυτό. Ψηφίζουμε την 412. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται λοιπόν. ΦΕΜ 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 419. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 420. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 426 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 429 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 432 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 433 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 436 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 438 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 439 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 440 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 77 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβα... Συμβιβαστική 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 47 υπέρ κατά αποχές Έμπλη 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 464 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 98 υπέρ κατά εποχές. Συμβαστική, συγγνώμη, 71. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 457 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 458 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 460 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 461 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 462 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 464 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 465 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 468 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 474 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 477 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 478 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 479 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 480 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 481 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ Β, Β, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 40, ε, συγγνώμη, 44, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 46, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ, ορίστε,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 κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία που θα γίνει ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Που. Geschlossen. Πέραση ψηφοφορίας. 27 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Αλλά πολλά ευχαριστώ και στους σκιώδεις εισηγητές και στην γραμματέα για την υποστήριξη. Την Άννα συγκεκριμένα θέλω να ευχαριστήσω. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. κυρία Φερχάιεν, για την πολύ καλά δομημένη και γρήγορη ψηφοφορία. Ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο, γιατί τα πήγε περίφημα. Ναι, κάνω την μπορώ, λέει Πρόεδρος. Ωραία. Περνάμε λοιπόν τώρα στην έκθεση πρωτοβουλίας διαρθρωτική και δημοσιονομική φραγμή στην πρόσβαση των πολιτισμού ο Μπόγκνταν Στρογεύσκη ήταν συγητή μα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε κύριε συγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να πω κάτι για να μπορέσετε και εσείς να πάρετε μια ανάσα, Πρόεδρε. Αυτή είναι η πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εξετάζουμε μία έκθεση που αφορά ολόκληρο το ζήτημα της πρόσβασης στον πολιτισμό. Βασίζεται στα δεδομένα του Βροβαρομέτρου και της Eurostat και θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό που βοήθησε στην κατάρτιση αυτής της έκθεσης, γιατί αυτά τα δεδομένα είναι πάρα πολύ ακριβή και αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο στον τομέα του πολιτισμού. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη δική μου ομάδα και τη Ιουστίνα γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε λοιπόν αφήσαμε στην ψηφοφορία. Ξεκινούμε με την τροπολογία 38, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 47. Πέραση ψηφοφορία. 15 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Έχουμε μια προφορική τροπολογία επίσης. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα ελέγξουμε την 65 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 13 υπέρ 14 κατά απορρίφθηκε συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 74 με προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται θα ελέγξουμε όμως ε, για να είμαστε σίγουροι 82 ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 11 προς 12. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 τρία τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε το τρίτο τμήμα της 103 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Η ισοψηφία 12 όλα. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίντ. Α, συγγνώμη, λέει πρόεδρος. Ήταν δύο τα τμήματα. Ξανά από Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πρώτο τμήμα. Δεν ήταν σαφές. Πέρας ψηφοφορίας. Όχι. Καλά. Ήταν 25 υπέρ και κανείς κατά. Τέλος πάντων. Τα έχασα. Δεύτερο τμήμα. Το πρώτο εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 108 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 111 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 114 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 δύο τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά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 137 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 139, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 140 ψήφι υπέρ,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 εγκρίνεται 33 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξουν. Το δεύτερο τμήμα της 33. Die Abstimmung ist eröffnet. Άρχεται ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία, 9 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο όμως. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές, απο... Ε, μάλλον δεκτό. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτό. 37 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Ποχές εγκρίνεται 4 υπέρ. Κατά. Ποχές εγκρίνεται 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 27 ψήφοι υπέρ, ομόφωνα δεκτή και συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Και τους και να συγχαρώ και να ευχαριστήσω, όπως φυσικά και τη γραμματεία. Μάλιστα. Προχωρούμε. Έκθεση πρωτοβουλίας για μία έκθεση εφαρμογής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία με εισηγήτρια την Ιντερ Γκαρθία Θάμπαλ. Ρουμπιά θέλεις το λόγο να πεις κάτι Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα για να μην καθυστερήσουμε τις ψηφορίες. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες για την καλή συνεργασία. Νομίζω ότι φτάσαμε σε συμβαστικές τροπολογίες που βελτιώνουν κατά πολύ την έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως την ομάδα μου που καθοδήγησε όλη αυτή την εργασία. Με την έκθεση αυτή νομίζω ότι όχι μόνο κάνουμε μια καλή αξιολόγηση για τη στρατηγική νεολαία, αλλά θέτουμε και τις βάσεις ε, για να πούμε στην Κομισιόν προς τα που θέλουμε να πάει στην επόμενη πρόταση που θα καταθέσει για τη στρατηγική περί νεολαίας. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Έντερ. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Ξεκινούμε με την τροπολογία 51. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές πραγματικά δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Να ελέγξουμε λοιπόν την 61 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, τώρα καταλαβαίνω όμως ότι είναι ξεκαθαρό. Ναι, πράγματι 22 κατά ήταν 5 υπέρ. Βοηθάει να σηκώνετε τα χέρια. 62 υπέρ κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Έμπλε 11 υπέρ. Α, όχι. Την 63. 63 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Πηγαίνω στροπολογία 68 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. αποχέ. απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75. Α, ναι, έχει αποσυρθεί. 76, 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, εντάξει, να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 76, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με συγχωρείτε γιατί όντως απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 18 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε,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 αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 109 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε την 110, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 17 ψήφοι υπέρ, εγκρίνεται λοιπόν. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, εκα... αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 115 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ευχαριστώ. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 115. Πέρασε. Απορρίπτεται. Μπορούμε να ξαναψηφίσουμε λοιπόν πρώτο τμήμα της 115. Πέρας. Εγκρίνεται, μάλιστα. Το πρώτο τμήμα λοιπόν εγκρίνεται, το δεύτερο απορρίπτεται. Περνάμε στην έμπλη 1, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη 22, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη 5, όχι. Ε, 117, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά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 Πού είμαστε? Α, στην 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 39. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 147. Πέρας. Απορρίπτεται. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MP37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ωραία. Βλέπω κουράζεστε, σαν να φαίνεται. 164. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η ισοψηφία απορρίπτεται. Ναι, αυτό πράγματι είναι κάτι που δεν μπορείς να δεις με το μάτι. Έμπλη 33, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, ας το ελέγξουμε. 170 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ. Α, με συγχωρείτε λέει πρόεδρος. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε την 198. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συγχωρείτε λοιπόν. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω ας το ελέγξουμε όμως ψηφίζουμε την 203 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 204 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 20 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Έμπλη 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλη ε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλη F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλη Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη C υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Οι 13 και οι 14 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία, ας ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίσουμε την 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. MPJ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ μη υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται θα το ελέγξουμε όμως να είμαστε σίγουροι έμπλ μη άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Έμπι νη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 23. 24, Entschuldigung, 24. Beschlossen? Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 1. Α, θέλετε να ελέγξουμε την 26. Ωραία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ξέρω πως είμαστε κουρασμένοι, όμως έχουμε κι άλλο. Έμπι γιώτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμπλη, D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε. Πέρας. Mit 14 zu 14 abgelehnt. Ισοψηφία 14-14 απορρίπτεται. Έμπλ L υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43. Περνάμε στην άλλη σελίδα. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47. Ας ελέγξουμε τη 45, άρχεται η ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά.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 Πέρας. 26 ψήφοι υπέρ, καμία κατά μία αποχή, τεράστια πλειοψηφία. Εγκρίνεται λοιπόν σχεδόν ομόφωνα. Συγχαρι... Συγχαρητήρια για την εισηγήτρια, για τους σκιώδεις εισηγητές, τους ε, υπαλλήλους γραμματείας και όλους τους συνεργάτες. Περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα, η οποία δεν είναι τόσο μεγάλη. Θα τα καταφέρουμε. Ελάτε, μια τελευταία προσπάθεια σχέδιο γνωμοδότησης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η εισηγητής είναι ο κύριος Τζαμπάτσκι. Θα θέλατε το λόγο? Όχι. Περνάμε λοιπόν αμέσως στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 και 41 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλω να βλέπω τα χέρια σας θα με βοηθούσε. Όχι μόνο τους συντονιστές, όλους. 63 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε την 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Α, την 69 ψηφίζουμε, λέει η πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Η 77 απορρίφθηκε, γι' αυτό και Περνάμε είναι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 και 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ Α, με διορθώνετε. Έχετε δίκιο. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε τη 12 άρχεται η ψηφοφορία Πέραση ψηφοφορίας 11 υπέρ 14 κατά απορρίπτεται 115 115 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ελέγχουμε την 115 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 14 προς 11 116 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε συγγνώμη αλλά 123 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 13 υπέρ, 12 κατά. Εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε παρακαλώ τη 13 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας 13 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ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 απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ α συγγνώμη έχει αποσυρθεί 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία η ονομαστική άρχεται Πέρας 20 ψήφι πέρα Καμία ψήφος κατά, πέντε αποχές εγκρίνεται, λοιπόν συγχαίρουμε και τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές και τη γραμματεία. Das war